Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ήρθαμε όλοι. Ξεκινάμε με πολύ μικρή καθυστέρηση και σας ευχαριστώ που ήρθατε εγκαίρως. Για τους γεωργούς, 9 ε, η ώρα ήταν ήδη η ώρα για το δεύτερο πρωινό, όχι το πρώτο. Άγρια χαράματα ξύπνουσαν οι άνθρωποι, οπότε 9 για, για τους γεωργούς παλιά ήταν και αργά. Περνάμε σε πολύ σημαντική και αρκετά δύσκολη ψηφοφορία για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, το Omnibus, το κανονισμό Omnibus. Θα ήθελα να μας κάνουν την εισαγωγή οι συγητές μας, ο κύριος Δες και ο κύριος Δεκάστρο, εγώ ε, να τονίσω ότι είναι σημαντικό γιατί όλες οι, ψηφοφορίες, όλες οι τροπολογίες που θα υπερψηφίσουμε σήμερα θα γίνουν ε, απευθείας δεκτές από τις αρμόδιες κατουσίαν επιτροπές. Θα κανονίσει η γραμματεία την περαιτέρω διαδικασία. Έγινε μια κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτροπή προπολογισμών και των άλλων συνδεδεμένων επιτροπών μεταξύ άλλων και τη δικιά μα. Είναι σημαντικό γιατί οι σημερινέ τροπολογίε θα πάνε κατευθείαν σε αρμόδιες επιτροπές. Ο κύριο Ντέ πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, που συνέβαλαν στο να καταρτιστεί αυτή η έκθεση. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδης ηγητές, ε, τον κύριο δεκάστρο τη διοίκηση. Ε, ευχαριστώ τους ε, συνεργάτες μου στην ε, πολιτική ομάδα και στο Προεδρείο, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε πάρα πολλά. Η Επιτροπή Προπολογισμών έχει πάντα επιφυλάξει κατά πόσον εμεί στην Επιτροπή Γεωργία θα ψηφίσουμε στην ώρα μα έγκαιρα. Και πρέπει να του πω ότι εμεί ε, τα καταφέραμε, τα ψηφίσουμε, ενώ η Επιτροπή Προπολογισμών ανέβαλε την ψηφοφορία. Εμεί λοιπόν ε, στην Επιτροπή Γεωργία εργαστήκαμε αποτελεσματικά και τα καταφέρνουμε στην ώρα μα. Θα ήθελα να πω στο μέλη τη πολιτική ομάδα ότι στο 104 ψηφίζουμε συν. Στον κατάλογο ψηφοφορίας απευθύνομαι στα μέλη της πολιτικής μου ομάδας ε, στο σημείο 104 θα υπερψηφίσουμε. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω και ελπίζω να έχουμε μια καλή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να πω ότι και εγώ θα ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τη γραμματεία, αλλά όχι εκ των προτέρων όπως έκανε ο εισηγητής, εγώ μετά το πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, πέραμε στην ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία, 99 του κυρίου Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104 που μας ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ντες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος ε, πιστεύω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 105, έρχεται η ψηφοφορία if this one is not adopted. Oh, yes, yes, yes, yes. yes. Okay. Przyjęta. Engrinete. We change place. Καλύτερα να αλλάξουμε θέσεις. Okej. Poprawka 105. O, sorry. We change. Poprawka 105. Η 105 εγκρίθηκε, οπότε η τροπολογία 2 καταπίπτει. Περνάμε στην 106. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 107. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 108 δεν την ψηφίζουμε γιατί εκρίθη μη παραδεκτή. Σας ε, το εξήγησε ο γραμματέας τον κύριο Φλάναγκαν. Περνάμε στην 109. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 111. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 117 και 118 μαζί για την επανομοιότυπη υπέρ εγκρίνονται. Τροπολογία 8 του κυρίου Δεκάστρου. Α, προηγουμένω όμως να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τις τροπολογίες 117 και 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 124 υπέρ. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 125. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 126 αργότερα. 127 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131. 131. Καπούτο και σάνι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 128. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά απορρίπτεται 135 υπέρ κατά απορρίπτεται 136 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 136 άρχεται Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 9 και 134. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 137 και 146 που είναι επανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 147, 145 μαζί. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνονται. 138. 38 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται έχουμε τώρα ένα σύνολο πανομοιότυπων τροπολογιών 139 και υπόλοιπε υπέρ εγκρίνονται 140 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 212... Ε, Ποιο Ποιος είναι υπέρ, 212. 212 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία δίστασα κάπως εγώ. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 212, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 181 αποσύρεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφόρια Εγκρίνεται και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή η συμβαστική τροπολογία, οπότε περνάμε στην τροπολογία 213 του κυρίου Δεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 213, άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ είδα ότι εγκρίνεται. Τέλος ψηφοφορίας και όντως εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 214. ή μάλλον όχι. 215 και 216. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογίες 217 και 218. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 219. Υπέρ. Εγκρίνεται. 220. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 220. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 221. Ποιο είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο? Όχι, δεν χρειάζεται. Ή μάλλον καλύτερα να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 24. Άρχεται ψηφοφορία. Εγώ είπα ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Εγώ το είχα πει και προηγουμένως ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 223 της κυρίας Σένερα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 224 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 225. Ή μάλλον όχι. 228 και 230 παρόμοιες υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 229 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 231. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 231. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται με μικρή διαφορά 2.32 και 2.33 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται τροπολογία 25 υπέρ εγκρίνεται 234 υπέρ εγκρίνεται 236 υπέρ εγκρίνεται περνάμε 239 ε, του κυρίου Γιάρη Περ. 239 Γιάρη Περ. Εγκρίνεται. 31. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. «238. Ποιος είναι υπέρ» «Εγκρίνεται» «237 υπέρ» «Κατά» «Απορρίπτεται» Πέντε τροπολογίες της κυρίας καλνιέται μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 2.42. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 33 και οι υπόλοιπες παρόμοιες υπέρ. Εγκρίνονται. 2.51. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 254 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 34 υπέρ όχι δεν χρειάζεται 253 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 256 υπέρ κατά απορρίπτεται 258 και 259, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 260 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος όμως προηγουμένως για τις τροπολογίες 258 και 259. Άρχεται η ψηφοφορία, μια και το ζητήσατε. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτονται. 260. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 381 ε, και 261 πανομοιότυπες υπέρ. Εγκρίνονται. 262. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 265. Όχι. Καταπίπτει. 35. 35 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 264. Καταπίπτει. 36. 36 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 266 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 267 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την προηγούμενη, την 266, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 266. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 267. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 267 απορρίπτεται. Η ίδια διαφορά ε, με τη 266 την οποία ελέγξαμε και ηλεκτρονικά. Πάμε στην 406. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 406. Άρχεται η ψηφοφορία. 406. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τροπολογία 405. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 407. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ε, 2.78. 2.78. 2,78 Ποιο είναι υπέρ είναι της κυρίας Καλνιέτη η τροπολογία εγκρίνεται ...274... ή μάλλον όχι... ...277... ...ποιος είναι υπέρ... ...κατά... Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 277. Άρχεται η ψηφοφορία. Διαδικαστικό ο κύριος Ντες. Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου μόλις μου επισήμαναν ότι δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα για την ψηφορία της τροπολογίας 267. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα της ψηφορίας. Κάτι δεν ακούσαμε καλά και από τη διερμηνία. Τη 267 την ψηφίσαμε ηλεκτρονικά και 267 θεώρησα ότι ήταν ίδια, το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά θέλετε να την ψηφίσουμε και τη 267. 267. Εντάξει, να ψηφίσουμε τη 267. 260. Εντάξει, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 267, αφού το ζητήσατε. Κανένα πρόβλημα, άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 267. 267. Otwieram głosowanie. Otwieram... Άρχεται η ψηφοφορία για την 267. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 38 του κυρίου Δεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 30 ή μάλλον 270. 270 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 293. Ποιος είναι υπέρ της 293, κατά. Καταπίπτει. Δεν, χρειάστηκε να Δεν χρειαζόταν να ψηφίσουμε. Πάμε στην 294 της κυρίας Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Ελεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 294 της κυρίας Νόιχλ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 295 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 296. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 297. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 297. Το ζήτησε η κυρία Γκυλερά, Άρχεται ψηφοφορία. 297. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά μόνο. 298. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγώ θεωρώ ότι εγκρίνεται με την ίδια διαφορά, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία για τη 298. Τέλος ψηφοφορίας. Όχι, απορρίπτεται. 299. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 300. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 303 της κυρίας Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ? 303. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 303. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 304. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 305 και 306 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 307 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 307. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 308 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 311 ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογίες 43 και 310 υπέρ, εγκρίνονται. 44 και 312 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. 313. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Εγκρίνεται. 46 ε, υπέρ. Εγκρίνεται. 314 υπέρ. Εγκρίνεται. 316. Ποιος είναι υπέρ. 316 υπέρ κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 347, 47 ε, συγγνώμη, ε, υπέρ, εγκρίνεται. 404. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 48. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 317 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 318 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 319 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία ηλεκτρονικός έλεγχος για την 319. άρχιτη ψηφοφορία. 319. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Εγκρίνεται. 320 υπέρ. Εγκρίνεται. 321 εγκρίνεται. 322 υπέρ. Εγκρίνεται. 323 υπέρ. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Εγκρίνεται. 326. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Εγκρίνεται. 346 υπέρ. Εγκρίνεται. 300 πρώτα όμως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 346 άρχεται η ψηφοφορία αυτό ζήτησε η Ομίγυρη τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Ευχαριστώ για την πρόταση ελέγχου. Περνάμε στην 327 του κυρίου Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 327. Γιατί ο κύριος δεν σήκωσε το χέρι του. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 54, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και η συμβαστική τροπολογία 9. Περνάμε στην τροπολογία 391. Περάσαμε μια-δυο σελίδες στον κατάλογο ψηφοφορίας. 391 του κυρίου Ντες. Ποιος είναι υπέρ της 391, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 394 της κυρίας Εράνς και άλλων. Ποιος είναι υπέρ της 394. Εγκρίνεται. Επειδή εγκρίναμε την 391, περνάμε κατευθείαν στην 394. Έτσι προβλέπει ο κατάλογος ψηφοφορίας. Η 394 εγκρίνεται, οπότε περνάμε στην 399. 391 του κύριο Ερντός. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 403 αποσύρεται. 55 του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Εγκρίνεται. 57 υπέρ εγκρίνεται. Ε, κύριε Νόιχλ, βλέπω, κουνάει το κεφάλι, αρνητικά, κάτι σας ενόχλησε, διαφωνείτε με κάτι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί 389 και 390 δεν έχουν πρόσημο. Οι 390 και οι 389 οι 390 και οι 389 δεν έχουν κανένα, καμία σημείωση δίπλα ότι καταπίπτουν. Γιατί λοιπόν δεν ψηφίζουμε για αυτέ. Είναι δύο τροπολογίε δικέ μου, δεν έχουν καταπέσει, ω εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε από αυτόν. Γιατί αν δεν ισχύει αυτό που λέω, τότε δεν ισχύει και ο κατάλογο ψηφοφορία. Κατά τη γνώμη τη γραμματεία. Επειδή εγκρίναμε την 391, θα πρέπει να περάσουμε κατευθείαν στην 394, έτσι λέει. Αν εγκριθεί 391, πάτε στην 394. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση της γραμματείας. Μια και εγκρίθηκε 391, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τις ενδιάμεσες. Πάμε κατευθείαν στην 394, η οποία επίσης εγκρίθηκε στο μεταξύ. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 468, αλλά στο μεταξύ θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά κάποιες άλλες τροπολογίες. Ξεκινάμε από την 428 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 428. Άρχεται η ψηφοφορία για την 428. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 435. Ποιος είναι υπέρ. 435. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 436. Ή μάλλον... Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε κατευθείαν στην 468. Ποιος είναι υπέρ της 468 τροπολογίας. Τον Δεκάστρο Ντόρφμα και Λαβία. Ποιος είναι υπέρ. 468. Εγκρίθηκε η προηγούμενη, οπότε πάμε στην 468. Δεν χρειάστηκε να ψηφίσουμε την 435. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 435. Καλό, σας ψηφίσουμε πρώτα διανατάσεις χειρός. 435, κατά. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 468 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Δεκάστρο Λαβία Ντόρφμαν. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 468. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 11 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ε, μία ψήφος διαφορά δεν θα επηρεάζει το αποτέλεσμα ούτως ή άλλως συνεννοούνται η κυρία Νόχλη με τον κύριο Καπούτο. Τελείωσε, τελείωσε η διαβούλευση. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 11 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 453. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 14. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 13. Ωραία ακολουθία. Πρώτα 14 και μετά 13. Τέλος πάντων, άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 13. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 458. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 74. Ποιος είναι υπέρ της 74. Εγκρίνεται και αυτή. 493 ναι 493 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται και αυτή 465 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 465 θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο ωραία άρχεται η ψηφοφορία για την 465 Ας μην προεξοφλώ το αποτέλεσμα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 462 τώρα. 462. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Εβδομήντα και 494 Ποιος είναι υπέρ κατά, μάλλον 474 και 479, συγγνώμη, ε, παρόμοιες, απορρίπτονται. 85 τώρα, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 88. Αλλά πρώτα να ψηφίσουμε την 501. Ποιος είναι υπέρ της 501. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα η 88 του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Ποιος είναι υπέρ. 93 υπέρ. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 93. Δεν ξέρω γιατί το ζητάτε. Εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 93. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγγνώμη κυρία μου, συγγνώμη κυρία μου. Εγκρίνεται, εγκρίνεται τελικά. Οριακά. 94. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 503. Υπέρ. Εγκρίνεται. 95 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κύριε Καπού, το δική σας είναι. Κατά. Απορρίπτεται. 97. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και 98 υπέρ. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Ο κύριος Ντεκάστρο βγάζει και φωτογραφία το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια, εγκρίνεται. Ε, συγχαίρουμε τους ε, εισηγητές της γνωμοδότησης. Φαντάζομαι τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριος Καπούτο, μια και στην αρχή έδωσε το λόγο στον ε, κύριο Ντες. Ο κύριος Δεκάστρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλά και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί πραγματικά έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτή η τελική ψηφοφορία αποδεικνύει ότι η δική μας επιτροπή σε τελική ανάλυση ήταν συμπαγής. Πράγματι πρόκειται για πολύ σημαντικές διατάξεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και ίσως και να είναι και η μόνη νομοθετική πράξη σε αυτή την ε, θητεία του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι να ακολουθήσουν οι τριμερείς διαλογοί διάλογοι με επιτυχία και αν δεν συμβεί και αυτό, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που ψηφίσαμε σήμερα να ενταχθεί στην μελλοντική νομοθεσία για την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε τους συγγητές μας, να τους συγχαρούμε. Αλλά δεν ολοκληρώσαμε ακόμη το έργο μας και δεν εννοώ το διάλογο Ε, μην ξεχνάτε ότι θα ξανάρθουμε στο θέμα του Omnibus. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύντομο κείμενο 3-5 σελίδες με σχόλια για το τι έγινε δεκτό, προς ποια κατεύθυνση βαίνει η Επιτροπή για να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε ε, στους συνομιλητές μας και να έχουμε την ενιαία γραμμή της Επιτροπής Γεωργίας. Ε, ναι, συγκαταβατικά και ο κύριος ε, Δεκάστρο, φαίνεται ότι συμφωνεί και ο κύριος Ντες. Ε, θα μας βοηθήσει πολύ ένα τέτοιο σύντομο κείμενο με, την, ε, το γενικό προσανατολισμό της Επιτροπής Γεωργίας. Ετοιμάστε το παρακαλώ οι συνεισηγητές. Θα είναι πολύ χρήσιμο για τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, για τους υπόλοιπους που δεν έχουμε παρακολουθήσει τόσο στενά όσο εσείς το θέμα. Ένα σύντομο κείμενο, το πολύ πέντε σελίδες, για να έχουμε συμπαγή τη θέση της Επιτροπής. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, ε, τις δεσμευτικές αιτήσεις μειώσει εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ο συντάκτης γνωμοδότης είναι ο κύριος Καπούτο Ήρθε η ώρα σας κύριε Καπούτο. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές για αυτή την έκθεση, γιατί πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη έκθεση και είναι και τεχνικής φύσεως. Ε, στις πολιτικές ομάδες υπήρχαν τρεις συγκεκριμένε ομάδες που ασχολήθηκαν με το θέμα. Δίσταντο οι απόψεις. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε τελικά σε μια θέση με την ψηφοφορία η οποία θα διαφυλάξει τα συμφέροντα του τομέα μας. Σας ευχαριστώ. Υπήρξε μεγάλη διάσταση απόψεων, όχι μεταξύ μόνο των πολιτικών ομάδων, αλλά και εντός των ομάδων υπήρχαν διαφορές. Το θέμα είναι να εξυπηρετήσουμε με τη θέση μας και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του γεωργικού κλάδου. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Πρώτα, τροπολογία 64. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Η 64 έγινε δεκτή, αλλά αφού επιμένετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ας το κάνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 64, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, γιατί εγώ έχω συν Αλμπερτ εδώ. Μήπως είναι λάθος ο κατάλογός μου. Όχι, ο εισηγητής εκπονεί τον κατάλογο ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορία οριακά. Ε, φαντάζομαι ότι θα με ευχαριστήσει ο κύριος Καπούτο, συντάκτης γνωμοδότησης. Εγώ είχα λάθος, λάθος α, α, ανέγνωσα τον κατάλογο και ψήφισε υπέρ. Πάμε στην 65. Ποιος είναι υπέρ? κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά απορρίπτεται. 68 οκτώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Εγκρίνεται. 75. 75. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά απορρίπτεται 77 υπέρ εγκρίνεται 78 αλλά πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 77 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 78. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 80 και 81. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 80... 85. Ποιος είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται 86 υπέρ εγκρίνεται 87 και 88 υπέρ κατά απορρίπτονται 89 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 89. Άρχεται ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Ποιος είναι υπέρ? Α, Μάλλον πάμε κατευθείαν στο 91 και μάλιστα στο δεύτερο τμήμα της 91. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98 της κυρίας Κέστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99. Η μελλονπρώτα πρώτα ηλεκτρονικός έλεγχος για την 98 της κυρίας Κέστιγκερ. Άρχεται η ψηφοφορία. 98 άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Κυρία Νόιχλου. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε την 5. Η τροπολογία υπερθυμών 5, το αποτέλεσμα δεν ήταν σαφές για την τροπολογία υπερθυμών 5. Καλώ Καλώς. Μια ναι, και μας το ζητάει η κυρία Νόιχλ, θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 5 που είναι του εισηγητού του κυρίου Καπούτο. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 5 του εισηγητού. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πριν αυτό είχαμε πει και περάσαμε στο δεύτερο τμήμα της 91 μετά από την 5. Και τώρα που είμαστε... 100. Τροπολόγια 100. Ποιος είναι υπέρ της κυρίας Νόιχλ και του κυρίου Μπράνεν. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι ίδια διαφορά, ίδιο αποτέλεσμα, άρα απορρίπτεται, αλλά θέλετε ας το, το εξακριβώσουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 101, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7 και 105 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 106. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 107 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις τροπολογίες 8 και 108. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 109. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 110. Ποιος είναι υπέρ? εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 και πάλι του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 11 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117 της κυρίας Γκέρλινγκ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 12 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 122. Για αρκεντές. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 13 του κυρίου Κάρθη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 της κυρίας Χόιμπουχ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά απορρίπτεται 19 υπέρ δεν χρειάζεται πάμε στην τροπολογία 1 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 1 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται και περάμε στην τροπολογία 23 του κυρίου Άγνιου. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 της κυρίας Κέστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται αλλά στο το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 26 άρχεται η ψηφοφορία απορρίπτεται τροπολογία 27 28. Ποιος είναι υπέρ της 28 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 42 υπέρ κατά απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32 άρχεται ψηφοφορία για την 32 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ? Υπέρ. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Εγκρίνεται. 30, 35 μάλλον. Υπέρ. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Εγκρίνεται. 39 ΔΕΣ και Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 39. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί κάποιος από τους ε, συντάκτες δεν ψήφισε την ίδια την τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 39 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 40. Ποιος είναι υπέρ. Μάλλον περνάμε στη 41 του κυρίου Φλάναγκαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 42. Κάρθη. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 3. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψυχοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Κέστιγκερ. Ή μάλλον 49 διορθώνει ο πρόεδρος. 49. Κέστιγκερ. Και πάλι ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 55 του κυρίου Κάρθη. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 5. και πάμε στην ψηφοφορία της τροπολογίας 62 των κυρίων Ντες και Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Καπούτο. Θέλετε μήπως στο λόγο. Απλά για να πω και πάλι τις ευχαριστίες μου για όλους και ας ελπίσουμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Να, και εμείς ευχαριστούμε. Αλλά θα μπορούσατε και εσείς να μας ετοιμάσετε κάποια σχόλια, δύο-τρεις σελίδες, σύντομο έγγραφο δύο-τριών σελίδων με τη θέση της Επιτροπής για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και στην επικοινωνία που θα έχουμε με τους ψηφοφόρους μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Συγχαρητήρια κύριε Καπούτο. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Την ψηφοφορία της γραμμοδότησης του κυρίου Σεράου Σάντος για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ειδικότητα του κυρίου Σάντος μεταξύ άλλων. Φαντάζομαι θα θέλετε το λόγο κύριε Σεράου Σάντος. Πολύ ευχαρίστω. Σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είχα σκοπό να ζητήσω το λόγο. Εν περιπτώσει, ευχαριστώ που μου τον δώσατε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό άρθρο του, της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συνοχή και την ανάπτυξη στις, στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Πρόκειται για γνωμοδότηση αυτή που συνέταξα εγώ γιατί αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, τις γραμματείες των δύο ε, επιτροπών για την ε, συνδρομή τους και επίσης να, ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις πολύ σημαντικές προτάσεις τους καθώς και τους και ηγητές για τις πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις τους. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε εισηγητά. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία, ξεκινώντας από τις τροπολογίες του κυρίου Νταντά, 7 τον αριθμό. Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Μαζί όλες και τις 7 του κυρίου Νταντά. Η κυρία Σάρα δεν συμφωνεί, οπότε ψηφίζουμε ξεχωριστά. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ, μια και η πλειοψηφία των ομάδων ήταν υπέρ της δέσμης, εν πάση περιπτώσει 7 υπέρ, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 10 της κυρίας Ριμπέιρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. 11 του κυρίου Φλάναγκαν. Τέλος ψηφοφορίας. Μάλλον εγκρίνεται να δούμε. ναι, ναι εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα για την τροπολογία 15, γιατί το ζήτησαν μερικοί. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15 έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. 17. Εγκρίνεται. Παρακαλώ τους συντονιστές ε, να δίνουν τις ενδείξεις και να σηκώνουν τα χέρια τους υπόλοιποι. 19 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, εγκρίνεται. 22. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 20... Όχι, 21 καταπίπτει. Οπότε πάμε στη συμβαστική τροπολογία α. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 24 υπέρ εγκρίνεται 25 υπέρ εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία Β άρχεται η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική τροπολογία σ Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στη συμβαστική D, γιατί εγκρίθηκε και η C. Συμβαστική D, άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 48 του κυρίου Νέκοφ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά απορρίπτεται 52 υπέρ εγκρίνεται 53 υπέρ κατά απορρίπτεται 54 υπέρ εγκρίνεται 55 υπέρ κατά απορρίπτεται 56 υπέρ ή μάλλον Καταπίπτει. Δεν ψηφίζουμε την 56, έχει καταπέσει, γιατί εγκρίθηκε η 48. Περνάμε στην 57, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 58 υπέρ, εγκρίνεται. 59 υπέρ, εγκρίνεται. 60 υπέρ, εγκρίνεται 61 υπέρ εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 30 ε, Μαΐου θα ψηφίσει η αρμόδια Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα πάει στην ε, Ολομέλεια του Ιουλίου. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ναι, απλώς για να ευχαριστήσω ε, όσους συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης που πραγματικά προωθεί τη συνοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τονίσει τη σημασία του προγράμματος για την ανάπτυξη πέθρου σε αυτές τις περιοχές. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Ε, σε λίγο θα περάσουμε στο σημείο 11, σε 5 λεπτά. 5 λεπτή διακοπή, γιατί ήταν πολύ εντατική η ψηφοφορία. Περιμένουμε στο μεταξύ και τους εμπειρογνώμονές μας, τους καλεσμένους μας. Πεντάλεπτη διακοπή και σε πέντε λεπτά συνεχίζουμε.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Θα σας πρότεινα να συνεχίσουμε τώρα, γιατί παρατείναμε την πεντάλεπτη διακόπη σχεδόν σε τέταρτο. Και ελπίζω θα, ότι θα επιστρέψουν και άλλοι ευρωβουλευτές μετά την εισαγωγή μου, ώστε να ακούσουμε τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες. Περνάμε στο σημείο 11, την παρουσίαση της ε, μελέτης που ζητήσαμε με θέμα την υποστήριξη ε, για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας ή τη στήριξη πολιτικής για την παραγωγικότητα έναντι της βιωσιμότητας της γεωργίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης γεωργίας και της πράσινης ανάπτυξης. Θέλουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα, αλλά να προωθήσουμε ταυτόχρονα και την πράσινη ανάπτυξη στην Γεωργία, τη φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη. Ένας όμιλος ανέλαβε τη μελέτη αυτή με την συμμετοχή τριών φορέων από το κλάδο της γεωργικής έρευνας και οικονομίας στην Ιταλία, από το Πανεπιστήμιο Βάγκενιγκεν των κάτω χωρών για την οικονομική έρευνα και από το ε, τμήμα γεωργικής οικονομίας του κέντρου Leibniz της Γερμανίας. Το θεματικό τμήμα Β ανέλαβε τη διαχείριση αυτής της μελέτης. Γι' αυτό και ευχαριστούμε θερμά αυτό το θεματικό τμήμα γιατί μας επέτρεψε να λάβουμε και στο παρελθόν πολύ εμπεριστατωμένες ε, θεματικές εκθέσεις και μελέτες με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να μας παρουσιάσει τους, τις βασικές τάσεις ε, της συνολικής παραγωγής, συντελεστών παραγωγής ε, στις τελευταίες δεκαετίες. Για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των πόρων και ταυτόχρονα τα, τους περιορισμούς, ε, τα, τα κριτήρια της ε, βιωσιμότητας. Αυτό γίνεται με την ανάλυση των επιμέρους πολιτικών ε, σε νομοθετικό επίπεδο προκειμένου να συμφιλιώσουμε την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα και να προωθήσουμε κάποιες συστάσεις για την πράσινη ανάπτυξη καθώς και ενός γεωργικού κλάδου που θα αξιοποιεί αποδοτικά τους σπόρους, θα είναι παραγωγικός, φιλοπεριβαλλοντικός και ανθεκτικός. Είναι μεγάλες προκλήσεις και μεγάλη επιβολή στόχη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω εδώ τους εμπειρογνώμονές μας, την κυρία Αναλίζα Τζέτζα και τον κύριο Ρομπέρτο Χένκε από το Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Οικονομίας της Ιταλίας που θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη τους. Πρώτα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας και θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Γεωργίας. Οι εμπειρογνώμονές μας έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά, μπορούν να τα κατανείμουν μεταξύ τους όπως θέλουν και να αποφασίσουν και με ποια σειρά θα μιλήσουν. Αυτά από πλευράς μου Παρακαλώ. Ίσως πρώτα η κυρία, η κυρία Τζέτζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόνο εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα κάνω την ε, παρουσίαση. Ε, παρότι βέβαια με τον ε, Ρομπέρτο συνεργαστήκαμε για αυτή τη μελέτη και ο Ρομπέρτο μπορεί να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβουλίο και την Επιτροπή Γεωργίας που μας ανέθεσε αυτή τη μελέτη και θα την παρουσιάσουμε σήμερα. έχει την εξή δομή η ομιλία μας. Ε, θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα τα οποία βασίζονται σε τρία θέματα. Στην ανάλυση των τάσεων, στην ανάλυση της ε, συνολικής παραγωγικότητας συντελεστών παραγωγής ε, και των πηγών που υπάρχουν στη Γεωργία. Κατόπιν θα γίνει η αξιολόγηση των εργαλείων γεωργικής πολιτικής και όχι μόνον αυτών και θα αναφερθούμε και σε κάποιες ε, μελέτες ε, περιπτώσεων και θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ε, συστάσεις. Όπως είπατε και εσείς, ο στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση της παραγωγικότητας των συντελεστών και των πηγών για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μία βιώσιμη εντατικοποίηση. Ε, μία από τις παραδοχές ε, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε στη μελέτη μας είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για την αξιολόγηση της ε, γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται για μια γενικότερη αξιολόγηση πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τελικά την πορεία της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας χρησιμοποίησαμε ένα πλαίσιο για την ανάλυση της ε, παραγωγικότητας, ένα πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει να μοιράσουμε την αύξηση της παραγωγής ε, σε διάφορους παράγοντες, ε, κυρίως στην αύξηση της αρρώσιμης επιφάνειας και των καλλιεργιών. Όσον αφορά το δεύτερο, πρόκειται για την ε, βελτίωση της ε, παραγωγικότητας ε, με βάση τους τεχνικούς παράγοντες και πρόκειται κυρίως για την αύξηση των εισρών, των inputs. Έχουμε λοιπόν την εντατικοποίηση, τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι αυτή, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί έχουμε παράγοντες οι οποίοι και αυτοί συνδέονται με διαφορετικές πολιτικές. Πολιτικές έρευνας, πρόκειται για την έγκριση παραγόντων όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, οι τιμές. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη δεν εξετάζουμε το θέμα των τιμών και της ανταγωνιστικότητας, παρότι είναι σαφές ότι και αυτό το στοιχείο είναι καθοριστική σημασία για να ορίσουμε τη δυναμική της γεωργίας. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την μπλε γραμμή η οποία δείχνει μακροπρόθεσμα την πορεία της αύξησης της παραγωγής. Βλέπουμε ότι η γεωργική παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διατηρήσει ε, θετικό πρόσημο, παρουσιάζει αύξηση, αλλά με την πάρο των ετών μειώνεται κατά τη αυτή η αύξηση. Αυτό λοιπόν οφείλεται, αυτή η μείωση οφείλεται και στη μείωση των ε, μοβ ε, στυλών που βλέπετε, ενώ παράλληλα διαπιστώνουμε την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας συντελεστών παραγωγής. Η γαλάζια στήλη είναι αυτή η ε, συνολική παραγωγικότητα. Οι κόκκινες στήλες δείχνουν την επιφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι την πάρδο των ετών μειώνεται η παραγωγικότητα η οποία προέρχεται από τις επιφάνειες αναφέρομαι στην πράσινη μικρή στήλη. Αν όμως ε, θέλουμε να δούμε τι ακριβώς ε, έγινε στα κράτη-μέλη, θα διαπιστώσουμε το αποτέλεσμα ποικίλει. Αυτό που βλέπουμε σε αυτήν την ε, διαφάνεια είναι μεσοσταθμικά τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπουμε την διαφοροποίηση του τι συνέβη τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη, ε, κυρίως αναπεριοχή. Έχουμε τα κράτη-μέλη του Βορρά, ε, κατόπιν ε, τις χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης η παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται και προέρχεται κυρίως από την αύξηση της παραγωγικότητας. Στις χώρες όμως της Νότιας Ευρώπης έχουμε αρνητικό ρυθμό παραγωγικότητας. Ε, αυτό το βλέπετε και στην πιο σκούρα ε, στήλη. Εκεί ε, βλέπουμε την παραγωγικότητα, διότι οι παράγοντες που υπήρξαν στις χώρες αυτές δεν ήταν επαρκείς έτσι ώστε να εξισορροπήσουν, να αντισταθμίσουν την απώλεια γης. Η πορτοκαλί στήλη δείχνει ότι υπάρχει μείωση της ε, παραγωγής ανά εκτάριο. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουμε αρνητική εξέλιξη της ε, παραγωγής διότι η μείωση της επιφάνειας ε, και της χρήσης των παραγόντων παραγωγής αυτό δεν μπόρεσε να αντισταθμιστεί από την αντίστοιχη πορεία της παραγωγικότητας. Εξάλλου, Βλέπουμε αυτή την εξέλιξη και με διάφορες άλλες μεταβλητές οι οποίες αφορούν τόσο την παραγωγικότητα των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούν στη Γεωργία για να κατανοήσουμε ε, πώς ακριβώς εξελίχθηκαν και ανακούληθησαν την ίδια πορεία η ε, βιωσιμότητα και η παραγωγικότητα πρέπει να δούμε κάποια ε, χαρακτηριστικά τα οποία θα εξετάσουμε και με περισσότερες λεπτομέρειες. Σε αυτό εδώ το γράφημα που είναι αρκετά περίπλοκο όμως ε, βλέπουμε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ε, συσχετίζεται με την παραγωγικότητα του άνθρακα. Και αυτό εξετάζεται και με την παραγωγή άνθρακα, ε, σε μετρημένη παραγωγή σε τόνους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι χώρες ε, στο πρώτο τετραγωνίδιο, ε, δεξιά αναφέρομαι, στο πάνω κομμάτι δεξιά του γραφήματος, οι χώρες ε, είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Δανία, η Ουγγαρία και εκεί διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής και παράλληλα μείωση των εκπομπών. Δηλαδή είναι χώρες οι οποίες κάτω από αυτό το πρίσμα είναι χώρες όπου διαπιστώθηκε βιώσιμη εντατικοποίηση. Αντίθετα, πάλι στο επάνω τετραγωδίνο, αλλά αριστερά έχουμε την Ουταλία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την ε, Ελβετία εκεί διαπιστώνουμε ότι μειώνονται οι εκπομπές. Αυτό όμως οφείλεται και σε μία μείωση της παραγωγής. Άρα δηλαδή η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα, τουλάχιστον με βάση αυτή τη μεταβλητή, ε, εκεί διαπιστώθηκε ότι υπήρξε κάποια εξισορρόπηση. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τις απόλυτες τιμές ε, και διαπιστώνουμε ότι όσον αφορά την παραγωγικότητα με μεταβλητή τον άνθρακα ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας ως ε, ε, πλεόνασμα αζότου. Αυτό στο κάτω τετραγωνίδιο δεξιά. Και εδώ Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, σε αυτές τις χώρες ε, η παραγωγή αυξήθηκε και μειώθηκαν οι εκπομπές αζότων εκτάριο. Άρα παραγωγικότητα και βιωσιμότητα ακολούθησαν την ίδια ακριβώς πορεία. Ενώ Αυστρία, Βουλγαρία, Πολωνία, εκεί διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής, όμως παράλληλα διαπιστώθηκε και αύξηση του πλεονάσματος αζότου. Και εδώ βλέπουμε τις απόλυτες τιμές αύξησης ε, του αζότου ανεκτάριου και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση κατά την πάροδο των ετών μέχρι και το 2014, αλλά τα απόλυτα επίπεδα είναι διαφορετικά, ποικίλουν, άρα δηλαδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικές προτεραιότητες στα κράτη-μέλη. Θελήσαμε λοιπόν να συσχετίσουμε ε, την πορεία της παραγωγικότητας ε, και της βιωσιμότητας με κάποιες ε, μεταβλητές οι οποίες μεταβλητές μπορούν να εκφράσουν πολιτικές ή διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της γεωργίας. Εξετάσαμε την εξέλιξη των δαπανών για την έρευνα στη γεωργία. Σε απόλυτες τιμές οι δαπάνες, οι επενδύσεις αν θέλετε, οι εθνικές επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη στη Γεωργία μειώθηκαν στη Δανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και αυξήθηκαν σε άλλες χώρες, ε, κυρίως ε, στις χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Όμως βλέπουμε εδώ τις δύο στήλες που δείχνουν τις δαπάνες σε ευρώ αν κάτοικο και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τελείως διαφορετικό απόλυτο επίπεδο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά τον αριθμό των πράσινων διπλωμάτων ευρεστεχνίας, αυξήθηκε ο απόλυτος αριθμός και αυτό οφείλεται κυρίως στην χρήση των υδάτων και στην διαχείριση των αποβλήτων. Όσον αφορά τώρα το φορολογικό καθεστώ για την έρευνα και την ανάπτυξη και εκεί υπάρχουν πολλέ ε, μεγάλες διαφορές στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχουν φορολογικά μέτρα για να ε, δώσουν όθηση στην καινοτομία. Έχουμε κίνητρα γενναιόδωρα, πούμε στη Γαλλία για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην περίπτωση της Γαλλίας και της ε, Ολλανδίας έχουμε νέους ε, γεωργούς οι οποίοι συστήνουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλες διαφορές στις ε, πολιτικές, τις περιβαλλοντικές, παραδείγματος χάνει στη χρήση των εργαλείων της αγοράς. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε το καθάριστο εθνικό προϊόν όσον αφορά στη γεωργία. Αυτό βέβαια δεν χρησιμοποιείται πολύ ω στοιχείο στην, ε, στην γεωργία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, διαπιστώσει κανείς την προέλευση και είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό το εργαλείο. Όμως ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για προγράμματα που έχουν σχέση με, με την εφαρμογή μέτρων για τα ζυζανιοκτώνα. Σε ορισμένες λοιπόν χώρες γίνεται επίσης ε, γίνεται χρήση και άλλων εργαλείων που δεν έχουν σχέση με την αγορά και εδώ λοιπόν έχουμε διαφορετικές παρεμβάσεις στα κράτη-μέλη. Ε, Παράδειγμα, είναι Λουά ε, Γκρενέλ στη Γαλλία, είναι ένα άλλο πρόγραμμα Origin Green στην Ολλανδία. Έχουμε και μια δανέζικη στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη ε, που έχει ως ε, βασικό στόχο τη διατήρηση το να παραμείνουν οι γεωργοί στη γη τους. Και στην Ολλανδία έχουν ληφθεί μέτρα που έχουν σχέση κυρίως με την χρήση των λοιπασμάτων. Στην έκθεση τη δική μας ε, έχουμε διαπιστώσει υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ε, όπως η ηλικία των γεωργών, ε, η ενημέρωση. Αυτά ποικίλουν στα κράτη-μέλη. Ε, λυπάμαι που δεν μπορείτε να δείτε καλά αυτόν τον πίνακα, όμως θέλω να πω το εξής. Αν δούμε λιγάκι το σύνολο των στοιχείων, θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι εμείς καταλήξαμε στο ότι υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την κατάρτιση, την ε, ανανέωση των γενεών. Όλα αυτά είναι ε, σημαντικοί παράγοντες ε, έτσι ώστε να προκύψει και να προκληθεί και καινοτομία. Εμείς εντοπίσαμε κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία, όπου εκεί υπάρχει μια θετική τάση στην αύξηση της ε, παραγωγής. Και αυτό εξηγείται από την αύξηση της ε, παραγωγικότητας, παράλληλα όμως μειώθηκαν και οι εκπομπές ε, θερμοκηπίου, του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ε, υπάρχουν πολλά κίνητρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία πράγματι κίνητρα αυτά έδωσαν όθηση στην εξέλιξη που σας ε, προανέφερα. Ε, υπάρχει, υπάρχουν επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οικονομικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με τις ε, Ισραήλ, οι οποίες όμως μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον. Μία άλλη ομάδα χωρών αφορά τις χώρες της Ανατολικής και της Ενότιας Ευρώπης. Η αύξηση της παραγωγικότητας, όπως σας είπα, εκεί δεν είναι επαρκής στις χώρες αυτές και ε, δεν αρκεί κυρίως για να αντισταθμιστεί η απώλεια γης. Έχουμε κάποιες, ε, κάποια βασικά συμπεράσματα για αυτό το πρώτο κομμάτι της έρευνας. Διεπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου πράγματι υπάρχει επιτυχία στο θέμα της ε, βιώσιμης εντατικοποίησης. Υπάρχουν πολιτικές πέρα από την κοινή γεωργική πολιτική, οι οποίες πολιτικές κατά τη δική μας άποψη έχουν επηρεάσει τη θετική πορεία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνοχή. Αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για να ε, στεφτεί από επιτυχία η στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης. Αν δούμε λιγάκι την κοινή γεωργική πολιτική, ε, θα θέλαμε να αναλύσουμε κάποια στοιχεία. Καταρχήν, ε, την γενικότερη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Είναι η βιώσιμη παραγωγή και οι ε, συνεργασίες για την καινοτομία. Σε αυτή τη διαφάνεια ε, χρησιμοποίησαμε τρία στοιχεία όπως και στο πρώτο κομμάτι. Βλέπουμε την εξέλιξη της ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής στο πάνω κομμάτι και στο κάτω κομμάτι βλέπουμε την εξέλιξη των μεταβλητών που είναι υγιή, ε, χρήση των ισρών και επιπτώσεις ε, από τις εκπομπές ε, του, του των, των φαινομένων θερμοκηπίου. Βλέπουμε λοιπόν την αύξηση της παραγωγής που είναι σταθερή, αλλά βλέπουμε και κάποια διαφοροποίηση και αυτό οφείλεται σε έναν από τους παράγοντες που έχουν σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στις εκπομπές. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής βοήθησαν στο να επιτευχθεί συνολικά ο στόχος που είναι να βελτιωθεί η παραγωγή και με βιώσιμο τρόπο. Ενώ λοιπόν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης αυτό δεν μπορούμε να το δούμε στο γράφημα η τάση σχετικά με την παραγωγή παρέμεινε αρκετά σταθερή. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η μία είναι μέχρι την εποχή Fisher, Μαξέρι μέχρι Fisher. Εκεί βλέπουμε την ε, μείωση της ε, παραγωγής ανάμεσα στην μεταρρύθμιση Fisher και στην μεταγενέστερη περίοδο υπήρξε και κάποια διαφοροποίηση, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της ε, παραγωγικότητας. Μείωση των διαφορών εισρώων και επίσης μείωση και της γεωργικής παραγωγής. Μετά το Health check υπήρξε συνεχής αύξηση της απόδοσης ε, και της παραγωγής ε, του άνθρακα. Άρα δηλαδή μείωση των εκπομπών. Αυτές οι τάσεις, όπως είπα και προηγουμένως, είναι λιγάκι συγκεχημένες, κυρίως όσον αφορά τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αν αναλύσουμε με λεπτομέρειες τα διάφορα εργαλεία της ΠΑΚ, πράγμα το οποίο κάναμε εμείς, θα διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μία μετάβαση προς ε, εργαλεία τα οποία εμείς ορίζουμε win-win, εργαλεία δηλαδή τα οποία μας επιτρέπουν να συμφιλιώσουμε την παραγωγικότητα με τη βιωσιμότητα. Όσον αφορά στο στόχο της βιώσιμης παραγωγής διαπιστώνουμε, έχουμε ένα στοιχείο το οποίο, ε, στο οποίο αντικατοπτρίζονται διάφορα εργαλεία και όσον αφορά αυτά τα εργαλεία εμείς αναλύσαμε την εθνική στρατηγική ε, κυρίως στα προκυπευτικά και στην Ιταλία. Η εθνική στρατηγική για τα οποροκυπευτικά, η στρατηγική αυτή είχε ως βασικό στόχο να αυξηθεί η δύναμη, η αγορά γενικότερα, έτσι ώστε να αυξηθούν κυρίως η οικονομική, να αυξηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν τα στοιχεία του ελέγχου και κατέστη απόλυτα σαφές ότι το εργαλείο αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας. Στην μελέτη μας επίσης διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων, οι επενδύσεις αυτές ε, έγιναν έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα καθεστώς ποιότητας ε, νοτιοανατολικά της Ιταλίας. Αυτό αφορά κυρίως το 78% της παραγωγής. Ως εκ τούτου διαπιστώσαμε ότι είχαμε αύξηση των εκτάσεων αλλά και της παραγωγής και επίσης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε αύξηση και της ε, συμμετοχής σε τέσσερα καθεστώτα ποιότητας, βιολογικές ε, καλλιέργειες, εθελοντισμός, ολοκληρωμένη παραγωγή και άλλου είδους πιστοποίησης. Εξάλλου, αναλύσαμε και κάποια άλλα αδύναμα θα έλεγα στοιχεία, ποια μπορεί να είναι αυτά τα αδύναμα στοιχεία και οι δικές μας συστάσεις αφορούν κυρίως την ενίσχυση του ρόλου που μπορούν να παίξουν στην αγορά οι οργανώσεις παραγωγών. Ε, πρέπει να στηριχτούν οι διαδικασίες ε, καινοτομίας ε, και εσωτερικοποίησης ε, μέσα από την εκπαίδευση των διαχειριστών των οργανώσεων παραγωγής. Να υπάρξει μια απλούστευση των ε, διοικητικών διαδικασιών. Απολύτως απαραίτητο. Ε, εξάλλου, καταλήγουμε και σε μια άλλη σύσταση που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά αφορά και άλλους τομείς ε, πολιτική. Αναφέρομαι στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για να μειωθούν ε, αθέμητες ε, πρακτικές, κυρίως στον τομέα των γεωργικών τροφίμων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι επ' αυτού υπήρξαν συγκεκριμένα συμπεράσματα μιας ομάδας υψηλού επίπεδου Μία ομάδα η οποία εργάστηκε μετά από ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο ελέγξαμε ήταν οι Ευρωπαϊκές Εταιρικές Σχέσεις για την Καινοτομία. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική φάση και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να εξετάσουμε μόνο τη δρομολόγηση και τον προγραμματισμό. Και νομίζω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. τουλάχιστον ε, όσον αφορά την ποσότητα. Αυτή η αρχική φάση αποδεικνύει ότι υπάρχουν και κάποια δύναμα σημεία τόσο σε ενωσιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Η δουλειά που έχει γίνει σε ενωσιακό επίπεδο ε, εστιάζεται κυρίως σε κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα, αλλά αυτό δεν διαδόθηκε επαρκώς. Πολλοί έχουν αναθεωρήσει το κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχουν προγράμματα τα οποία ε, ξεπερνούν τα εθνικά ή τα περιφερειακά όρια και αυτό για να μην υπάρχει επικάλυψη στις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται. Σε επίπεδο κρατών μελών. Πράγματι υπάρχει κάποια επικάλυψη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που διαπιστώθηκε είναι ότι είναι απαραίτητο να δοθούν περισσότερα κίνητρα ε, στη συμμετοχή ε, και στον χρόνο που απαιτείται ε, για να συμμετέχουν οι γεωργοί σε αυτές τις μορφές συνεργασίας. Ε, υπάρχουν ε, κάποιοι ενδιάμεσοι innovation brokers όπως αποκαλούνται οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους ε, γεωργούς σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Όσον αφορά λοιπόν στις διάφορες πολιτικές, ανακεφαλαιώνοντας, εμείς καταλήξαμε στο ότι υπήρξαν πράγματι αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική. Και στην έκθεσή μας αναφέρουμε επίσης ε, ότι οι μεταρρυθμίσεις, τα μέτρα είχαν επιπτώσεις, αλλά δεν ήταν οι προσδοκόμενες. Και αυτό οφείλεται και στο ότι υπήρξαν πάρα πολλές ε, εξαιρέσεις ε, στους κανόνες, εξαιρέσεις ε, οι οποίες τελικά οδήγησαν στο να υπάρχει υπερβολική ευελιξία στα κρατη όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά νομίζω επ' αυτού έχουν γίνει αναφορές και σε άλλες εκθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από άλλους εμπειρογνώμονες. Πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν εκμεταλλευτεί βέβαια και την ευελιξία αυτή που προσφέρθηκε για να υπάρχουν καλύτερες περιβαλλοντικέ επιπτώσεις από τις μεταρρυθμίσεις. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα μπορούσαν να έχουν πολύ θετικέ επιπτώσει, Αναφέρομαι κυρίω σε αυτά που έχουν σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή ή με την καινοτομία. Και η σύγχρονη σύγχρονες τεχνολογίες έχουν σίγουρα θετικές επιπτώσεις, δηλαδή μπορούν ε, να έχουμε πολλά θετικά μέτρα όπως είναι η τηλεανείχνευση, η χρήση των ρομπότες, στις ε, καλλιέργειες και στη γεωργία γενικότερα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε πράγματι μια βιώσιμη εντατικοποίηση στη γεωργία. τα, οι διοικητικές ε, διαδικασίες ε, ε, αυτές αποθαρρύνουν τους γεωργούς το να συμμετέχουν στα νέα προγράμματα και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί αυτό το γράφημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Αυτό που θα ήθελα απλά να δείτε είναι ότι εμείς κάναμε μελέτες ε, περιπτώσεων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη εντατικοποίηση σε επίπεδο ε, εταιρεία, επιχείρηση, σε επίπεδο εθνικό. Μέσα από όλα αυτά μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα οικονομικό προφίλ και να ε, εντοπίσουμε και τις πηγές και τους πόρους να καταλήξουμε στο τι συμβαίνει με τη χρήση της γης σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ε, προσεγγίσεις και εμείς, όπως σας είπα, ε, χρησιμοποίησαμε διάφορα παραδείγματα. Αυτά μπορούμε να τα συνενώσουμε σε μία και μόνο στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη είχαμε μελέτες ε, περιπτώσεων, πέντε ε, συγκεκριμένες ε, μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποίησαμε στις δικές μας τις μελέτες που έχουν, χρήση, έχουν σχέση με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Εμείς εξετάσαμε μια συγκεκριμένη περιφέρεια όπου έχουμε επιτυχημένες βιολογικές καλλιέργειες. Κάναμε μελέτες για ε, αρρώσιμες καλλιέργειες στην Ολλανδία, για τη χρήση των ε, ρομπότ ε, για την παραγωγή γάλακτος στην Ολλανδία, συγκεκριμένες πρακτικές για γεωργία ακρίβειας. Τελικά, πού καταλήξαμε με όλες αυτές τις μελέτες περιπτώσεων καταλήξαμε σε αυτά ε, που είχαμε δει και σε σχέση με τα συνολικά στοιχεία. Βλέπουμε ότι η καλύτερη διαχείριση, η έρευνα και η ανάπτυξη ε, μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα μπορούν να παρα... αυξάνονται και οι δύο παράλληλα, δηλαδή να μην υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. οι γεωργοί στο βαθμό που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν ε, βιώσιμες μορφές καλλιέργειας. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από το πλαίσιο πολιτικής, όπως επίσης ε, και από το ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια συνοχή αν θέλετε ανάμεσα στα διάφορα μέτρα. Οι γεωργοί τους οποίους εξετάσουμε στο πλαίσιο των περιπτώσεών μας δεν επιθυμούν να εκτεθούν σε νέους κινδύνους και γι' αυτό στις επιλογές τους ε, δεν ε, συμπεριλαμβάνουν πλήρως ε, και το περιβαλλοντικό στοιχείο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη ξικίωση με την περιβαλλοντική διάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας φαύλος κύκλος μπορεί να προκύψει για όλες τις δραστηριότητες, τις ανθρώπινες και πολιτικές δραστηριότητες γιατί βλέπουμε ότι πρόκειται εδώ για κοινέ αρχές, κοινέ προσεγγίσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει πράγματι να επιδιώκουμε την βιώσιμη καινοτομία. Και μόνον αυτό αλλά και την ανάπτυξη συστημάτων, αποτελεσματικών συστημάτων. Αυτά είναι καθοριστική σημασίας παράγοντε για να επιτύχουν πρωτοβουλίε σε τοπικό επίπεδο. Και τέλος υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων. Η ε, στρατηγική εντατικοποίησης, ε, βιώσιμης εντατικοποίησης, η στρατηγική αυτή προφανώς και χρειάζεται επενδύσεις για να υπάρξει κάποια αρχή και αυτό τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, όσο και σε επίπεδο υποδομών. Όταν δηλαδή μιλάμε για τις πρωτοβουλίες ε, χρήσης γης σε τοπικό επίπεδο. Θα τελειώσω την ομιλία μου με κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις. Η βιώσιμη εντατικοποίηση και η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι ξεκάθαρο στόχο στην κοινή γεωργική πολιτική. Ίσως λοιπόν απαραίτητο να γίνουν ξεκάθαρο στόχος έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογούμε καλύτερα τα εργαλεία που έχει η κοινή γεωργική πολιτική για να χρησιμοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία να υπάρχει και μία ολοκλήρωση, μία συνέχεια ανάμεσα στους στόχους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο στόχος ε, που είναι η βιώσιμη εντατικοποίηση. Να χρησιμοποιούνται εργαλεία ε, τα οποία καταλήγουν σε λύσεις ε, που ικανοποιούν όλους, win-win, Η αύξηση της ε, παραγωγικότητας και η αύξηση της βιωσιμότητας είναι δύο πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς ε, να τα επιτύχει την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Οι δικές μας οι αναλύσεις ε, μάλλον υπήρχε αυτή η παραδοχή κατά το παρελθόν. Όμω, εμεί αποδείξαμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό και αύξηση τη πραγματικότητα και τη βιωσιμότητα. Για να γίνει όμω αυτό, πρέπει να υπάρχουν απλουστεύσει και καλύτερη επικοινωνία. Επικοινωνία τόσο όσον αφορά του στόχου που επιθυμούμε να πετύχουμε, όσο και τα εργαλεία και τα αποτελέσματα τη έρευνα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει βελτιωμένος διάλογος ανάμεσα στην επιστήμη, την πολιτική, τους γεωργούς, τη βιομηχανία που παράγει τη νέα τεχνολογία. Η κυκλική γεωργία, κατά την άποψή μας, είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί που θα χρησιμοποιηθούν κατά τα επόμενα έτη για να ενισχυθούν οι δυνατότητες πράσινης ανάπτυξης στο γεωργικό τομέα. Και όσον αφορά αυτό, εμείς ζητάμε ή μάλλον βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο ε, να υπάρξει, να υπάρξει ε, περισσότερο η πράσινη διάσταση στην κοινή γεωρική πολιτική. Ελπίζω να παρέμεινα μέσα στο χρόνο που μου είχατε διαθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σε αυτή την ε, τελευταία διαφάνεια. βλέπετε και τα ονόματα των συνεργατών μας εγώ και ο συνάδελφός μου, ο κ. Χένκε, είμαστε από το Εθνικό Συμβούλιο για την Έρευνα ε, και την Οικονομία στην Ιταλία και οι δύο συμμετείχαμε σε αυτή την έρευνα που σας είπα, όπως και το Wagening Economic Research και το ΤΣΑΛΦ, ε, το Κέντρο ε, Γεωργικών Ερευνών που βρίσκεται στο Leibniz, στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Ζέτζα. Είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου σήμερα, γι' αυτό και σας ε, αφήσαμε χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Άλλωστε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτής της μελέτης. Γι' αυτό και έκανα σκόπιμο να μην σας διακόψω νωρίτερα. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε. Ως είδηση θα περάσουμε στη συζήτηση, γιατί το θέμα ήταν ιδιαίτερος ενδιαφέρον και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τέτοιου είδους μελέτες και έρευνες και ε, πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τους ε, συντάκτες αυτής τη μελέτης. Ο κύριος Δενανό πρώτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια μελέτη με πολλά και περίπλοκα και αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα θέματα. Περίπλοκα θέματα και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι είναι μια γεωργική πολιτική βιώσιμη. Εγώ αυτό που άκουσα με μεγάλη προσοχή είναι ότι βάλατε δίπλα-δίπλα δύο λέξεις την εντατικοποίηση και τη βιωσιμότητα. Δεν πρόκειται για σας για δύο λέξεις ε, οι οποίες ε, φαίνεται να είναι αντίθετες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εντατικοποιήσει και την ίδια ώρα να έχει ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Καταρχήν, όσον αφορά την έρευνα, τα αποτελέσματά σας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και φορέων, πώς τα συνδυάσατε. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών εδώ για τέτοιου είδους ε, έρευνες. Μιλήσατε επίσης για την φορολόγηση των παρασιτοκτόνων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω. Μία άλλη ερώτηση. Η μείωση της παραγωγικότητας μετά από την αποσύνδεση έτσι το παρουσιάζεται ότι υπάρχει σημαντική μείωση της παραγωγικότητας μετά από την αποσύνδεση, την αποσύζευξη. Η χρήση εδώ των βιοκαυσίμων και βάσει της οδηγίας και της τροποποίησης της οδηγίας για την ενέργεια που είχε επιπτώσεις όσον αφορά το βιοντίζελ και την εθανόλη. Έχετε λάβει υπόψη σας τις επιπτώσεις για το γεωργικό κόσμο όλων αυτών των ε, τροπολογιών, της οδηγίας παραδείγματος Θα ήθελα να μου δώσετε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ κυρία Ρανς Γκαρσία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη. Θα συνεχίσω όμως τα ισπανικά. Πραγματικά πολύ αξιόλογη η μελέτη σας με ενθουσίασε και την άκουσα με μεγάλη προσοχή, αλλά με παραξένεψε που παραλείψετε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ηλικία των γεωργών και την κατάρτιση των γεωργών. Γιατί μας ενδιαφέρει η μέση ηλικία των γεωργών στα κράτη-μέλη. Και η στάση που έχουν στα νέα συστήματα παραγωγής, στην καινοτομία, τις επενδύσεις. Και η κατάρτιση είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί κάποιος μπορεί να είναι πολύ νέος να μην έχει παρακολουθήσει κάποια προγράμματα κατάρτισης και άρα να μην είναι ιδιαίτερα δραστήριος και να μην μπορεί να αξιοποιεί τις νέες ευκαιρίες. Ε, από τη μεταρρύθμιση του Επιτρόπου Μαξάρη ε, μέχρι σήμερα μας ε, παρουσιάσετε κάποιες γενικές γραμμές, αλλά θα ήθελα μια πιο ενδελεχή μελέτη των συνεπειών. Και ε, αυτή η επινόησή μας για ενδιάμεσα αναθεωρήσεις των ε, πολιετών δημοσιονομικών πλαισιών, αυτό το έβριμά μας δημιουργεί μια βεβαιότητα στο γεωργικό κλάδο. Γιατί στο παρελθόν οι γεωργοί γνώριζαν ότι είχαν μια σταθερή περίοδο, μια σταθερή επταετία, κατά την οποία δεν θα άλλαζαν ε, οι προϋποθέσεις ή οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια όμως οι όροι αλλάζουν στα μέσα της περίοδου λόγω αυτού της επινόησης της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Οπότε στερείται τη σιγουριά πια ο Γεωργός γιατί γνωρίζει τα πρώτα δύο χρόνια τι θα συμβεί αλλά μετά από το τρίτο και μετά δημιουργείται μια βεβαιότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν φαίνεται αυτός ο αντίκτυπος κατά την ε, ε, επικαιροποίηση των ε, επενδύσεων ή των προσπαθειών που κάνουν για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και πρώτα απ' όλα την ανταγωνιστικότητά τους οι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σουλαζό. Oui, merci, Président. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα μοντέλο, το γαλλικό γεωργικό μοντέλο που είναι πραγματικά παραδειγματικό. Θα ήθελα να πω ότι πάνω απ' όλα πρόκειται για επιχειρηματίες, ανθρώπους που με μεγάλη συνείδηση σέβονται το περιβάλλον. Πρόκειται για άτομα με πολύ καλή κατάρτιση που γνωρίζουν τον τομέα τους και νομίζω ότι μπορούμε να διατηρήσουμε, να βελτιώσουμε την παραγωγή με έναν βιώσιμο τρόπο στη Γεωργία. Όσον αφορά τώρα την ε, τεχνολογία, η αρχή της ε, υγρομετρίας, δηλαδή ο βαθμός υγρασίας ε, στην ατμόσφαιρα, είναι κάτι που σαφώς λαμβάνεται υπόψη. Επίσης τα φυτοφάρμακα και όταν πρόκειται για φυτά που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η χρήση φυτοφαρμάκων 10, 20, 30% ίσως και παραπάνω όταν γίνεται μια σωστή αξιολόγηση και εδώ μπορεί ακόμα περισσότερο να βελτιωθεί ε, αυτό. Η βιωσιμότητα λοιπόν βεβαίως μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής. Αυτό είναι το συμπέρασμα νομίζω που μπορούμε να φτάσουμε. Κύριε Χόιμπους. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, αυτά που μας παρουσιάσατε. Σημειώσατε επίσης ότι υπάρχει μία αντίσταση, μία αμφιβολία των ίδιων των γεωργών όσον αφορά τις επενδύσεις. Διστάζουν δηλαδή να επενδύσουν. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία. Εγώ εδώ φαντάζομαι αυτό που είπατε, όσον αφορά την εντατικοποίηση, δηλαδή περισσότερες επενδύσεις για κάποιες ε, παραγωγές οι οποίες έχουν ε, κέρδος όταν διατεθούν τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Γιατί οι γεωργοί διστάζουν. Όταν μιλάμε για εντατικοποίηση, θα πρέπει να μην ε, ξεχνάμε ότι βεβαίως παράγουμε περισσότερο τα προϊόντα που μπορούν να πολιθούν στην αγορά. Άρα μιλάμε για εντατικοποίηση, περισσότερη παραγωγή και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι τα προϊόντα αυτά εάν δεν διατίθεται, δεν πολλούνται, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μιλάμε για εντατικοποίηση αν δεν υπάρχει αγορά που να μπορεί να απορροφήσει αυτά τα προϊόντα. Το θέμα τώρα της μέτρησης που κάνετε και της σύγκρισης με τις ε, εκπομπές. Βεβαίως υπάρχουν ε, τεχνολογίες ε, που αφορούν το περιβάλλον που θα πρέπει να αξιολογηθούν και να μετρηθούν. Αλλά όταν μιλάμε για εντατικοποίηση, θέλω να ξέρω και τις επιπτώσεις στη γη. Κοιτάμε δηλαδή και το έδαφος, τις επιπτώσεις στη γη ή εσείς έχετε λάβει υπόψη σας μόνο το θέμα των εκπομπών. Έχετε λάβει δηλαδή το θέμα και των επιπτώσεων στη γη. Ευχαριστώ κύριε Μπόκοβιτς. Ε, αυτά που μας ε, είπατε είναι ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Μπορεί κανείς να τα προγραμματίσει θαυμάσια για την ε, μελλοντική γεωρική πολιτική. Υπάρχουν όμως δύο αντιφατικά πράγματα. Αφενός έχουμε την βιωσιμότητα και την εντατικοποίηση, τα οποία ναι μεν αντιφατικά, αλλά μπορεί κανείς και να τα συνδυάσει. Με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και να επιτύχουμε και τη βιωσιμότητα. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη μελέτη που μας παρουσιάστε, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε ε, περισσότερες γνώσεις αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη ε, γεωργία και αν θέλουμε να έχουμε και μια κυκλική ε, γεωργία. Γιατί και η γεωργία κάπου και αυτή πρέπει να εντάσσεται γενικότερα μέσα στον κύκλο της οικονομίας. Αλλά ακούσαμε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γεωργία μετακινείται περισσότερο προς βορειοδυτική Ευρώπη. Μας δείξατε τα αποτελέσματα της παραγωγής ε, στα σχετικά γραφήματα και κατέστη σαφές ότι η Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ επιτυχημένη, τα πάει πολύ καλά στη γεωργία, βελτιώνεται η γεωργική παραγωγή σε αντίθεση με τη Νότια Ευρώπη ή με τις ε, χώρες μετάβασης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα πολύ προσεκτικά Βλέποντας ε, την ε, εντατικοποίηση, διαπιστώνουμε ότι η εντατικοποίηση είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο ε, στη Βόρεια σε αντίθεση με την Νότια και την Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οφείλουμε να στηρίζουμε τη βιώσιμη γεωργία, την ολοκληρωμένη προφανώς, αλλά παράλληλα πρέπει και να δημιουργούμε τις ε, προϋποθέσεις ε, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και σε χώρες ε, του Νότου ή σε αυτές που βρίσκονται σε φάση μετάβασης, όπως χαρακτηρίζονται. Εγώ έρχομαι από τη Σλοβενία και έχω διαπιστώσει το εξής. Πάρα πολλά μέτρα της κοινή γεωρικής πολιτικής είναι τόντι καλά. Όμως η παραγωγικότητα μειώνεται ριζικά και πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που κυριαρχεί δεν είναι το κέρδος, αλλά κυρίως το να καλλιεργούνται οι εκτάσεις. Εγώ λοιπόν στηρίζω αυτά που είπατε και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τη γεωργία ακριβίας, ε, νέες ε, σύγχρονες τεχνολογίες, όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην κοινή γεωργική πολιτική. Ε, χρειαζόμαστε μέτρα με τα οποία μπορούμε να προάγουμε την κινητικότητα στη γεωργία. Και επίσης ε, οφείλουμε να βελτιώσουμε και την, ε, τον συσχετισμό ανάμεσα στην παραγωγικότητα και τη ζήτηση. Σήμερα γίνεται λόγος και για τα ευφυή χωριά, τα smart villages. Αυτά τα χρειαζόμαστε για να προσελκύσουμε νέους γεωργούς και για να υπάρχει βιωσιμότητα στη γεωργία. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουμε προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει απευθείας πώληση τροφίμων. Σας συγχαίρω για τη μελέτη σας που δίνει πολύ καλές απαντήσεις και αυτές τις απαντήσεις θα πρέπει στο μέλλον να τις λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντική η μελέτη σας. Πολύ αξιόλογη. Και πραγματικά προσεγγίζετε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ ορθολογικό τρόπο. Και εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τομείς τους οποίους έχουν ε, προοδεύσει με διαφορετικούς ρυθμούς. Διαπίστωσε και πάλι ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το είπατε κι εσείς ότι μεταξύ, και νο... μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, ε, η κατάσταση των γεωργών διαφέρει αισθητά. Κάτι που δείχνει ότι είναι αδύνατο να έχουμε ομοιόμορφη κοινή γεωρική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε πραγματικά να λάβουμε υπόψη και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές. Γιατί οι διαφορές δεν υπάρχουν μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των περιφερειών στις ίδιες ε, χώρες. Επίσης είπατε ότι τα κράτη-εθνή έχουν ε, πολλές αρμοδιότητες για τη γεωργία, αλλά ίσως στο μέλλον θα πρέπει τέτοιου είδους αρμοδιότητες να τις ε, περιορίσουμε κάπως για να έχουμε κοινά αποτελέσματα. Μας ε, παρουσιάσετε κάποιους λόγους για αυτές τις διαφορές. Είπατε ότι στις ανατολικές χώρες μέλη τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα, η παραγωγικότητα έχει μειωθεί ενώ η μέση ηλικία των γεωργών αυξάνεται. Για ποιους λόγους όμως υπάρχουν αυτές οι διαφορές, γιατί αν δεν εντοπίσουμε τα αίτια του κακού δεν πρόκειται να διορθώσουμε την κατάσταση και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δεν αρκεί μια διάγνωση και διαπίστωση της κατάστασης. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις αιτίες αυτής της κατάστασης Μπορεί να μην προλάβατε λόγω του περιορισμού του χρόνου να μας παρουσιάσετε και τις αιτίε που ίσως στη μελέτη σας ε, τις εντοπίσατε και τις αναλύσατε. Αλλά θα μας ενδιαφέρει και αυτό το σημείο. Γιατί ε, και στις ε, νεότερες χώρες μέλη, στις χώρες Βαλτικής για παράδειγμα, οι γεωρικές ταπάνες είναι εξίσου υψηλές με αυτές της Ολλανδίας, για παράδειγμα παρόλο που η γεωργία μας ουσιαστικά αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 90. Μέχρι τότε η γεωργία δεν υπήρχε σχεδόν, ενώ στις ε, χώρες της Δυτικής Ευρώπης η παράδοση της γεωργίας είναι μακραίωνη και η πείρα πολύ πλούσια, ενώ η δική μας ε, γεωργία αναπτύχθηκε πριν από ε, λίγες δεκαετίες. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές. Επίσης, σωστά είπατε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ε, συμπράξεις καινοτομία ή τις εταιρικές σχέσεις της καινοτομίας και να έχουμε στοχευμένα προγράμματα ώστε να εξοικειωθούν ε, περισσότερο οι γεωργοί μας με την καινοτομία και τις ευκαιρίες ε, που προσφέρει. Να διδαχθούμε από τα παραδείγματα της Ολλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές και ανισότητες και στα γεωργικά εισοδήματα μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών της Ευρώπης. Ενώ οι δαπάνες είναι ε, περίπου παρόμοιες, τα γεωρικά εισοδήματα διαφέρουν και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, όπου οι γεωργοί έχουν χαμηλά εισοδήματα δεν έχουν δυνατότητα επενδύσεων, μια και δεν τους περισσεύει τίποτα για να επενδύσουν. Επίσης, η τιμή παραγωγής είναι, οι τιμέ στην παραγωγή είναι πολύ χαμηλότερε στις χώρες που έχουν πιο μακρά γεωργική παράδοση. Οπότε και η διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών είναι υψηλότερη και ο βαθμός οργάνωσης είναι πολύ ψηλό. Είναι μερικές φορές και 80%. Ενώ σε εμά ο βαθμός οργάνωσης των γεωργών είναι πολύ χαμηλό, 10-15%. Κάτι που αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική ισχύ των γεωργικών συνεταιρισμών που δεν μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές. Επίσης, δεν έχουμε, αρκετούς, ε, διακλα... Ε, δεν έχουμε αρκετές διακλαδικές οργανώσεις που θα συνεργάζονται με τους παραγωγούς και τους μεταποιητές και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατάρτιση και ενημέρωση των γεωργών. Επίσης, πριν από ένα-δύο χρόνια καταργήσαμε τις χαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Ε, ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου στην ύπεθρο, στην παραγωγικότητα της γεωργίας μας, κατά τη γνώμη σας. Και πώς επηρέασε αυτή την προσέλκυση των νέων γεωργών, γιατί αν εγώ θέλω να επενδύσω στη γεωργία, πρέπει να έχω μία ε, βεβαιότητα σε δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορώ να επενδύσω αν δεν είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρω να αποσβέσω τις επενδύσεις μου και να έχω και απόδοση αυτών. Θέλουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα και σιγουριά για να ενισχύσουμε τις γεωργικές επενδύσεις. Πολύ χρήσιμη μελέτη, ίσως θα πρέπει να την ε, γνωστοποιήσουμε σε ευρύτερου κύκλους και στα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί όχι, για να ενημερωθούν καλύτερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Σε ευχαριστώ. Δεν σας ε, περιόρισα στο χρόνο αγόρευσης, αλλά ε, μην κάνετε κατάχρηση, παρακαλώ. Η κυρία Γκυλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση της μελέτης που πραγματικά μας ε, εφοδίασε με πολύ χρήσιμα στοιχεία. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Στα συμπεράσματά σας αναφερθήκατε στην ανάγκη καλύτερου και πιο διευρυμένου διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να προσαρμόσουμε τα μέτρα της γεωργικής πολιτικής στους στόχους της και είπατε ότι χρειάζεται καλύτερος διάλογος μεταξύ ε, γεωργών, ε, πανεπιστημιακών, επιστημόνων, ε, πολιτικών και επιχειρηματιών. Γιατί έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι μερικοί έχουν το ρόλο του κακού και άλλοι το ρόλο του κακού σε αυτή την αλυσίδα. Θα ήθελα στις απαντήσεις σας να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων. Και δεύτερη ερώτηση. Μερικές φορές ζητούμε τη λήψη κάποιων μέτρων υπέρ της καινοτομία και της έρευνας, γιατί και η Γεωργία αλλά και ο κάθε τομέας που δεν επενδύει στην έρευνα και στην ανάπτυξη δεν έχει μέλλον. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια κοινωνική απόρριψη ή μια δυσπιστία ακόμη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο απέναντι στην καινοτομία γιατί έχουμε κάποια καινοτόμα μέτρα στον αγοραπιστιστικό τομέα που μερικές φορές προκαλούν προθυμία, δυσπιστία έως και απόθυση μερικές φορές, η απόρριψη της καινοτομίας. Και αυτό ίσως οφείλεται στην έλλειψη επιστημονικών γνώσεων. Και αυτό με ανησυχεί γιατί αναφυσβήτα θα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην έρευνα. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για να αποφεύγουμε τέτοιες, τέτοια απόρριψη, τέτοια απροθυμία της κοινωνίας, ακόμη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μερικές φορές κατά της καινοτομία ή νέων ευκαιριών που δίνει η έρευνα. Νομίζω ότι αυτή την απόρριψη και αυτή την αρνητικότητα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και ποιος ε, πώς θα μπορούσαν οι επιστήμονες να, ε, να εξηγήσουν καλύτερα την ανάγκη της καινοτομίας προς την κοινωνία, ώστε να γίνει πιο εύκολα δεκτή η ανάγκη αυτής της καινοτομίας. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να είμαι από την αρχή της παρουσίασής σας και ίσως κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί από αυτά που είπατε. Καταρχήν κατανοώ ότι υπάρχουν δύο επίπεδα. Υπάρχει η κατάσταση ως έχει, το status quo, με την παρούσα κατάσταση όπως έχει με τα κράτη-μέλη και την ίδια ώρα υπάρχει η εξέλιξη στο εσωτερικό ενός κρατους μέλους για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάπως δύσκολο μου φάνηκε να καταλάβω από αυτά που είπατε στη γραπτή σας παρουσίαση, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θετικά βήματα στο λεγόμενο status quo, αν δηλαδή συγκρίνει κανείς το ένα κράτος μέλος με ένα άλλο. Υπάρχει ένα κράτος μέλος που έχει καλύτερες επιδόσεις από ένα άλλο. Όμως δεν λέτε τίποτα όσον αφορά την ίδια χρονική περίοδο για τις επιδόσεις ενός κράτους μέλους. Αν παραδείγματο χάρη υπήρξε εξέλιξη περισσότερο σε κάποιον τομέα ή σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή την συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων τομέων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ότι η βάση εκκίνησης, αν θέλετε, οτι η βαση κίνηση, αν θελετε μπορει να μην είναι ίδια. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν συγκρίνουμε ακριβώς δύο παραδείγματος χάρη παρόμοια πράγματα ε, στην ίδια διαδικασία, στον ίδιο τομέα και στην ίδια χρονική περίοδο. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές από την, Επιτροπή Γεωργίας. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις και να παρουσιάσω κάποιες αμφιβολίες που έχω. Το πρόβλημα της αξιοποίησης των πιο φτωχών εδαφών και δυσκολίες της ε, ε, καλλιέργειάς τους. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι θα είχαμε πολύ περισσότερες ε, επενδύσεις σε αυτά τα πιο φτωχά εδάφη αν η αποδοτικότητά τους ήταν μεγαλύτερη. Οπότε, αν επενδύσουμε περισσότερο σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, θα τις βοηθήσουμε να επιβιώσουν πολύ πιο εύκολα, γιατί μερικές φορές σε αυτές τις ε, περιοχές που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες η επιβίωση είναι πολύ πιο δύσκολη. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Ξέρουμε ποια είναι η στρεματική απόδοση και πώς επηρεάζει την, ε, ε, την εντατικοποίηση. Ποιο είναι όμως το όριο της εντατικοποίησης στη γεωργία. Πού θα βάλουμε το όριο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύγκριση μεταξύ των ε, παλιότερων και των πιο νέων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια οι παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εποφελήθηκαν από την ΚΑΠ. Ενώ την, εποχή, την ίδια εποχή χώρες Ανατολικής Ευρώπης υπάγονταν στο σοσιαλιστικό καθεστώς. Κάτι που δημιουργήσε μια υστέρηση στην ε, γεωργική τους ανάπτυξη. μήπως ήταν πολύ πρόωρη η εφαρμογή των ίδιων ακριβώς εργαλείων και ε, στις χώρες της Ανατολικής και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ό,τι αφορά την ΚΑΠ. Γιατί οι συνθήκε είναι πολύ διαφορετικές στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και το κλίμα, οι μετεωρολογικές συνθήκες, ε, αλλά και η κατάσταση της γεωργίας ίδια είναι πολύ διαφορετική. Και είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές που αφισβητούμε το κατά πόσο είναι ε, εύκολο να αντιμετωπίσουμε με παρόμοιο τρόπο τις προκλήσεις να έχουμε τους ίδιους στόχους. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε μια διαφοροποίηση των μέσων και των εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών και να κρατήσουμε μια ακριβοδίκαιη προοπτική στην ε, κατανομή των ενισχύσεων. Πριν μίλησα για το που βάζουμε το όριο της εντατικοποίησης στη γεωργία. Αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το επίπεδο εντατικοποίησης επηρεάζει την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, πού είναι το όριο της βιώσιμης ανάπτυξης, από ποιο σημείο και μετά θα κρίνουμε μία ε, γεωργική ανάπτυξη ως βιώσιμη. Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτό το ποσοστό ή των δαπανών ε, ή της, των ισρών της γεωργίας για να κρίνουμε ότι η ανάπτυξη θεωρείται βιώσιμη, ότι η γεωργία είναι βιώσιμη. Επίσης, το θέμα των υδάτινων πόρων είναι σημαντικό συντελεστή ε, για τη Γεωργία. Προφανώ. Αυτό το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και λέμε ότι το νερό επηρεάζει και την ποιότητα των εδαφών, των γεωργικών εκτάσεων. Πολλές ε, χώρες ε, κρίνουν ότι το πρόβλημα των εδαφών είναι εθνικό και ότι δεν χρειάζεται παρακολούθηση των εδαφών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι όμως μια υπεκφυγή που προσπαθούν, που ε, χρησιμοποιούν μερικές χώρες. Γιατί μερικές φορές η αποκατάσταση του καλού επίπεδου ενό υποβαθμισμένου εδάφους απαιτεί πολλές δαπάνες και αυτό το αποφεύγουν δυστυχώς χώρες μέλη λόγω του ύψους των δαπανών που χρειάζονται. Αυτό δεν ξέρω μετά τις απαντήσεις αν προκύψουν και νέες ερωτήσεις και δεν ξέρω αν τις ε, νέες ενδεχομένως απορίες που θα έχουμε θα μπορούσαμε να σας τις στείλουμε και γραπτός για να μας απαντήσετε. Πάντως η μελέτη σας ε, είναι πολύ χρήσιμη και τώρα και στις μελλοντικές συζητήσεις ε, για την διαμόρφωση της ε, μελλοντική κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί είναι σημαντικό. Κάναμε κάποιες τέτοιες αναλύσεις και στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus και οι αναλύσεις αυτές θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Επίσης, είπαμε πόσο έχει αυξηθεί η γεωρική παραγωγή από τη δεκαετία του 50. Μερικές φορές ε, έχει πολλαπλασιαστεί και μερικές φορές τίνουμε να κατηγορούμε μόνο τους γεωργούς για την υπερβολική εντατικοποίηση και απαιτούμε παρόλα αυτά να κρατήσουν την παραγωγικότητά τους, αλλά υπάρχουν όρια και στην παραγωγικότητα που συνδέονται και με την ε, εντατικοποίηση της γεωργίας. Αυτό το θέμα θα το θέσω και στους συντονιστές. Ώστε στο μέλλον να ζητήσουμε μια ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και μια συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στη μελέτη σας. Και δεν το λέω αυτό για σήμερα, ε, το άμεσο μέλλον, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να επιληφθούν ε, οι συντονιστές και να ζητήσουν από τους αρμοδίους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να παρουσιάσουν σχετικές προτάσεις. Αυτά είχαμε, όπως είπα και πριν, την πολυτέλεια του χρόνου σήμερα, γι' αυτό επεκταθήκαμε κάπως στη συζήτηση. Ήρθε η ώρα να λάβετε και εσείς το λόγο. Έχουμε αρκετό χρόνο, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να τον εξαντλήσουμε και να τελειώσουμε στις 12.30. Δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσουμε και το τελευταίο λεπτό του χρόνου μας. Έχετε το λόγο πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ερωτήσεις και τις ε, παρατηρήσεις που κάνατε. Εγώ δεν θέλω προφανώς ε, να εξαντλήσω τα 45 λεπτά, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ένα θέμα το οποίο τέθη αφορά στην εντατικοποίηση. Τι είναι αυτή η εντατικοποίηση. Εμείς σας δείξαμε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο που χρησιμοποίησαμε για τις αναλύσεις μας η αύξηση της ε, παραγωγικότητας δεν συνδέεται μόνο με την ε, μεγαλύτερη χρήση παραγόντων, αλλά σχετίζεται κυρίως με την καλύτερη χρήση των παραγόντων ε, των συντελεστών παραγωγής. Μέσα από αυτό μπορούμε να επιτύχουμε την καινοτομία, να κάνουμε καλύτερη χρήση της εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη. Μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε αυτή τη βελτίωση. Άρα δηλαδή δεν πρόκειται για χρήση χημικών παραγόντων, σαφώς και όχι. Εμείς συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους και δηλαδή αυτά τα οποία αγοράζουν οι γεωργοί και ε, άλλοι παράγοντες που δεν έχουν σχέση με χρήμα αλλά έχουν σχέση με ε, κοινωνική ωφέλεια. Εμείς ε, σας καταδείξαμε δύο μόνο παράγοντες, δύο συντελεστές ε, ε, που έχουν σχέση με τη γεωργία. Σας καταδείξαμε το θέμα των εκπομπών, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως ο συντελεστής της ε, βιοπαραγωγής. Ε, στην έκθεση υπάρχει αυτός ο συντελεστής, μπορεί κανείς να τον δει. Ε, και επίσης αυτό που εξετάσαμε είναι και η εντατικοποίηση στη χρήση της γης. Η επιλογή των συντελεστών συνδέεται είτε γιατί είναι σημαντικοί οι συντελεστές αυτές για την πολιτική της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή αυτά τα οποία θεωρούμε ως προτεραιότητα, είτε διότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία μπορεί κανείς να συγκρίνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα δηλαδή και αυτό καθόρισε την επιλογή μας. Όσον αφορά στην ερώτηση σχετικά με την ηλικία και την εκπαίδευση των γεωργών, κοιτάξτε, στη σελίδα 30 της έκθεσής μας υπάρχουν όλα τα στοιχεία για την Ευρώπη. Δεν σας τα έδειξα σε διαφάνεια, αλλά εκεί μπορεί να βρείτε αυτά τα στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά την φορολόγηση των φυτοφαρμάκων, αυτό είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία υιοθέτησαν κάποια κράτη-μέλη. Ε, Βεβαίω, ε, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο αυτό στη Δανία και πολύ καλά και στη Γαλλία. Είναι πολιτικέ οι οποίε αναθεωρούνται, πρέπει να το πω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για την ίδια την ε, τεχνολογική εξέλιξη που χαρακτηρίζει τα φυτοφάρμακα, ε, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς ε, να βρει αυτή την ε, ευαίσθητη ισορροπία. Παραδείγματο χάνει. στη Γαλλία. Υπήρξαν επενδύσεις προς όφελος των γεωργών και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να μπορεί κανείς να λάβει μέτρα τα οποία συμβάλλουν στο να επιτρέψει την χάνεται βελτίωση της γεωργίας. Όσον αφορά τώρα στο θέμα των ε, βιοκαυσίμων ε, στο τέλος ε, αναφερόμαστε στην κυκλική οικονομία. Νομίζω ότι στην Ευρώπη ευτυχώς δεν γίνεται πια λόγος για παραγωγή εθανόλης από ε, γεωργικές καλλιέργειες πρώτης γενιάς. Ε, όμως ε, αυτό είναι στην αιχμή του δόρωτος ε, και σε σχέση με τα κατάλοιπα και την απόκτηση βιοενέργειας. είναι δηλαδή περιβαλλοντικά και τεχνολογικά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας επιτρέψουν να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την χρήση των πόρων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ολοκληρώσουμε και ένα κύκλο χρήσης των πόρων. Είπατε να υπάρχει περισσότερος διάλογος ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, ε, δηλαδή ανάμεσα στην έρευνα, την πολιτική και τους γεωργούς. Εγώ αναφέρθηκα στα focus groups. Ε, υπήρξε λοιπόν μεγάλη προσπάθεια να ε, συγκεντρώσουμε όλους αυτούς ε, που μπορούν να συνεισφέρουν, να τους συγκεντρώσουμε στις ε, Βρυξέλλες και από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα αυτής της ε, προσπάθειας δεν είχε απήχηση στις ομάδες των γεωργών διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θέλει κανείς να συζητήσει και γι' αυτό το λόγο τι γίνεται, ξεκινάμε από το μηδέν. Μεγαλύτερη λοιπόν ρευστότητα στο σύστημα και είναι σαφές ότι μιλάμε για ένα νέο καινοτόμο εργαλείο όμως ε, ένα στοιχείο το οποίο έχει ένα τεράστιο δυναμικό και διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Γεωργίας ε, έχει μια έκθεση η οποία σίγουρα θα είναι και πολύ πιο λεπτομερής από τη δική μας. Ίσως ο Ρομπέρτο θέλει να λάβει το λόγο να μιλήσει για την ε, κυνηγιουργική πολιτική. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια στοιχεία ε, που νομίζω ότι έχουν σημασία για την γεωργική πολιτική και τις ε, μεταρρυθμίσεις. Έγινε λόγος, παραδείγματο χάρη, για τις ε, συνεχείς αλλαγές οι οποίες λαμβάνουν χώρα και οι αλλαγές αυτές δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας για τους γεωργούς. Όμως αυτό είναι σημαντικό, πρέπει κανείς να κατανοήσει και τον αντίκτυπο των μέτρων. Σήμερα συζητάμε για τις μεταρρυθμίσεις μετά το 2020, ενώ όμως τρέχουν ακόμα οι παλιές. Ε, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε ακριβώς γνώση τον αντίκτυπο κάποιων εργαλείων, κυρίως των πλέον καινοτόμων εργαλείων στη γεωργία. Ε, είναι σαφές ότι υπάρχει έντονη διαφοροποίηση στη γεωργία στην Ευρώπη και διαφορετικός και ο αντίκτυπος. Δηλαδή έχουμε ολοκληρωμένες γεωργίες, ε, έχουμε και μορφές γεωργίας ε, που είναι πολύ περιφερειακές, ε, γίνονται από μικρούς γεωργούς, από πιο ηλικιωμένου ε, γεωργούς, επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την επόμενη γενιά. Άρα δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε τελικά ποιοι είναι οι αποδέκτες της καινοτομίας και κατά πόσον η καινοτομία πράγματι μπορεί να εισαχθεί σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων. Διότι σήμερα η γεωργία και οι λειτουργίες που αναπτύσσει ο γεωργός είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένες. Δηλαδή αναπτύσσουν σε επιχειρήσεις τους οι γεωργοί και άλλες λειτουργίες. Ως εκ τούτου ε, και η καινοτομία και στην καινοτομία θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια διαφοροποίηση. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα βασικά που ήθελα να προσθέσω και όσον αφορά τα εργαλεία της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής, Είπαμε ότι σήμερα η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί ε, μια βεντάλια εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχει ένας μεγάλος εμπλουτισμός της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε όχι ως μία πρόκληση, αλλά ως προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε να έχουμε εργαλεία τα οποία είναι πιο κοντά στη γεωργία και μας ε, επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε καλύτερα συνέργειες. Συνέργειες ανάμεσα σε εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα... Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν ε, παρεμβάσεις, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο. Ως εκ τούτου, ας ε, ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ε, ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες και αν έχετε καλοσύνη να μεταφέρετε και τις ευχαριστήσεις σας σε όλους τους ερευνητές. αν έχουμε άλλες ερωτήσεις θα σας τις υποβάλουμε σε γραπτή μορφή. Και ίσως μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ίσως βέβαια ε, να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα μέχρι το καλοκαίρι, αλλά ίσως από το Σεπτέμβριο μπορούμε να προβλέψουμε ε, μία ακρόαση. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω. Στα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι βλέπω και γι' αυτό λοιπόν κλείνουμε. Επόμενη συνεδρίαση, αν θυμάμαι καλά, στο Στρασβούργο. 15 Μαΐου νομίζω είναι Δευτέρα. Ε, φαντάζομαι ο κύριος Ντες θα μου στείλει παρατηρήσεις. Θα μου πει ότι δεν έχει νόημα να γίνεται συνεδριά στο Στρασβούλ Τι να κάνουμε. Δυστυχώς ε, έτσι είναι τα πράγματα. Και ε, ξέρετε, αν μου το πείτε θα το πω και εγώ ότι ναι, και σήμερα όμως που έγινε ακρόαση δεν ήσουν παρόν. Αυτά. Καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους. Ε, τελικά μπορέσαμε να συμπυκνώσουμε τις ε, εργασίες μας και ε, ως εκ τούτου δεν έχουμε συνεδρίαση για σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε έναν τριμερή διάλογο στις 3 ε, η ώρα, αλλά δεν θα έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής. Αυτά ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους Ιερμηνείς.